Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απάντησα στην τελευταία υποθέτω ερώτηση και δεν θα σας καθυστερήσω πολύ περισσότερο στα συμπεράσματά μου. Θέλω απλά να μοιραστώ μαζί σας ε, μια αίσθηση κατεπήγοντος θα έλεγα για την δουλειά που πρέπει να κάνουμε τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαι πεπισμένος ότι αν αποτύχουμε στα επόμενα δύο χρόνια να συνδεθούμε εκ νέου με τους πολίτες για τους οποίους βρισκόμαστε εδώ, τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή, τότε το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα απειληθεί εάν δεν συνδεθούμε εκ νέου με αυτούς που λέμε ότι εκπροσωπούμε. Τότε θα γυρίσουν την πλάτη τους ε, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και μάλιστα ο άνθρωπος την έφτιαξε καλά την Ευρώπη. Είναι ε, έλεγα η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα από τα καλύτερα προγράμματα και σχέδια ειρηνικής συνύπαρξης στον κόσμο. Και όταν λέω την έφτιαξαν ε, οι άνθρωποι εννοώ, δεν εννοώ άνδρες ή γυναίκες, Η γυναίκα μου άλλωστε λέει για να με πειράξει ότι όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, ο Θεός ήταν γυναίκα. Εν πάση περιπτώσει, η επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν μεγάλη και δεν θα πρέπει να πάμε πίσω, δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Και έχω την αίσθηση τα τελευταία χρόνια βλέποντας και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και η Ευρώπη σήμερα. Αυτή η τεράστια οικονομική κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη δεκαετία του 30, αυτή η ανυπόφορη αίσθηση απειλής από το εξωτερικό, είτε από τον υπερεθνικισμό της Ρωσίας, είτε από τον ακεραιοφρονισμό στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά δείχνουν δύσκολες στιγμές για πρώτη φορά μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι γονείς φοβούνται για το μέλλον των παιδιών τους. Δεν υπάρχουν εθνικές απαντήσεις σε αυτές τις απειλές και σε αυτή την αίσθηση. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή απάντηση. Πρέπει όμως για να το κάνουμε αυτό αποδεικνύοντας ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Ίσως να θεωρείτε ότι το χαρτοφυλάκι μου είναι τεχνικής φύσεως. Όμως το να υπάρξουν πιο θετικά και χρήσιμα αποτελέσματα σε επίπεδο νομοθετικό για τον Ευρωπαίο πολίτη είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξανασυνδεθούμε με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων το μέλλον είναι εν μέρη και στα χέρια μας. Πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε σωστά και σε υπηρετικό θα έλεγα επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο, σεβόμενος τις εθνικές διαστάσεις βέβαια, που συμπεριέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν δεν αλλάξουμε τη στάση μας ε, τα επόμενα χρόνια και αν δεν ε, καθορίσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας, οι οργανώσεις μας, οι οργανισμοί μας, ε, δεν θα έχουν και πάρα πολύ μεγάλο νόημα πια για τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτό δεν θα αφήσουμε να συμβεί, γιατί αν έχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό η Ευρώπη περισσότερο από όλες τις άλλες υπήρους είναι η δυνατότητα προσαρμογής στις νέες προκλήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα προσαρμοστούμε, θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και θα πούμε σε λίγα χρόνια στα παιδιά μας ότι σας δίνουμε την Ευρώπη σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι τη βρήκαμε πριν 10 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τιμεμάντς και για το ότι κρατήσατε το χρόνο σας. Τώρα, ε, τα μέλη της Επιτροπής της Διάσκεψης των Πρόεδρων που θα ε, κάνουν την αξιολόγηση. Ε, θα συναντούμε στις 6 ώρα.